Δεν μπορώ να Varmt välkomna till dagens ehm, Καλώς ήρθατε σε αυτή τη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Γυναικών. Να σας καλωσορίσω. Θα έχουμε γλωσσική αρρωγή από πλευρά των διερμηνών μας. Έχουμε επίσης και μια ομάδα επισκεπτών. Προέρχονται από το κόμμα της Εστεράς στο Έλσμποργκ Επιτροπή, Συμβούλιο αλλά έχουμε επισκέπτες και κάποιους ε, μεταφραστές της Επιτροπής που έχουν την έδρα του στο Λουξεμβούργο και ήρθαν εδώ για να δουν πώς δουλεύει το κοινοβούλιο. Όλοι, καλώς ορίσατε. Έχουμε δεδομένη την ε, μέσα διάταξη, δεν ξέρω αν υπάρχει καμία αίτηση για τροποποίηση. Όχι, επομένω θεωρώ ότι έχει εγκριθεί. Δεύτερο θέμα είναι οι ανακοινώσει τη Προέδρου. Σας υπενθυμίζω, συνάδελφοι, ότι αύριο πρόκειται να γιορτάσουμε τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας. Εδώ και ως ε, εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική θα πάμε στις 9 ε, η ώρα στο ημικύκλιο του αίθουσα της ε, Ολομέλειας. Θα γίνει μια δημοσία ακρόαση μέχρι τις 12.30. Το πρόγραμμα έχει διανεμηθεί και ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολλούς συναδέλφους που θα έρθουν στην ακρόαση η οποία έχει ως θέμα την βία κατά των γυναικών. Η σχετική καμπάνια του Κοινοβουλίου λέγεται «Μπορούμε να το σταματήσουμε». Επίσης, συνάδελφοι, πρέπει να σας ενημερώσω και για κάτι άλλο. Οι αντιπρόεδροι, αλλά και οι συντονιστές της Επιτροπής μας, θα έχουν γευμαργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής, όπως παραδοσιακά γίνεται, Ε, ευκαιρία του γιορτασμού αυτού. Και για φέτος αυτό έγινε στο Στρασβούργο. Κύριος Μπαρόσο, κυρία Ρέντινγκ, η κυρία Μάλμστρομ παρευρέθηκαν. συζητήσαμε τα θέματα της βία των γυναικών, τις μισθολογικές διαφορές, την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών. Αυτά που συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Τρίτο θέμα στη ημερησία διάταξη. Μπορούμε να αρχίσουμε να το συζητούμε. Γιατί αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Η συγγήτρια είναι η κυρία Λούλινγκ, η οποία επίσης παρίσταται. Για αυτό το θέμα δεν θα γίνει συζήτηση. Σήμερα θα γίνει στη συνεδρίαση της 20 Απριλίου. 8 Τετάρτου λίγη προθεσμία υποβολή τροπολογιών και 4 και 5 Μαΐου θα γίνει η ψηφοφορία. Οπότε και θα υποβληθεί κατά την ε, δεύτερη ολομέλεια του Μαΐου η έκθεση στην ε, ολομέλεια του σώματος. Και τώρα σκητάρει στην κυρία Λούλη για να μας πει δύο λόγια όσον αφορά το θέμα για το οποίο είναι η συγγήτρια. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σας πω ότι τελικά ολοκληρώθηκε η επίσημη εκδοχή για την κοινή θέση. Όπως αυτή παγιώθηκε τον Νοέμβριο στο Συμβούλιο. Πολύ πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό και καθυστέρησε και η δική μας διεκπαίδευση. Πάντως συνεργαστήκαμε και με τη γραμματεία, είδαμε και εκπροσώπους της Ισπανικής Προεδρίας, συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους της Σουηδικής Προεδρίας πριν την Ισπανική και όλα αυτά παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να σας πω ότι μου δημιουργεί κάποια συγκρατημένη ικανοποίηση η εκείνη αυτή θέση, μια που σε κάποια σημεία ε, υπάρχει πρόβλημα, δεν μας συμβαίνει μαζί μας το Συμβούλιο όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, την αποχρεωτική ασφάλιση. Ε, γιατί από αυτό το σημείο, από ό,τι φαίνεται, το Συμβούλιο δεν έχει περιθώρια λιγμών. Πάντως, ε, κατά τα λοιπά, ε, έχουμε περίπου 12 τροπολογίες με τις οποίες συμφώνησε το Συμβούλιο. Οπότε τον Απρίλιο ελπίζω οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν θα μας βοηθήσουν να πάμε σε δεύτερη ανάγνωση με ένα κείμενο το οποίο θα συγκεντρώνει την ε, συνένεση όλων των πλευρών ούτως ώστε όλο το θέμα να διεκπαιρεωθεί επί Ισπανικής Προεδρίας γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μην το πάμε και στην επόμενη Προεδρία και κυρίως άπαξ και αυτή είναι η βελγική προεδρία που δεν το θέλουμε για πολλού λόγους να γίνει κάτι τέτοιο. επομένω. πέρασε ένα χρόνο από τότε που άρχισε η πρώτη αναγνώση. Πήρε πολύ χρόνο, βλέπετε. Ε, γίνανε βήματα πρόοδου, μικρά, αλλά γίνανε. Τον Απρίλιο θα τα συζητήσουμε με το κείμενο το οποίο πρόκειται να σας διαβιβαστεί. Ευχαριστώ. Ο κύριο ε, Ρομέδο. Μια ερώτηση. Εάν κατάλαβα αυτά που μας είπατε, <clears throat> στην πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή των γυναικών για την κοινωνική ασφάλεια, η εισφορά τους. Εάν αυτό αληθεύει, σε ποιο πλαίσιο ε, προβάλλεται αυτό το επιχείρημα. Και αν ισχύει κάτι τέτοιο, και σε σχέση με τη θέση που εμεί έχουμε προασπιστεί πολλέ φορέ στο Ευρωκοινοβούλιο, διερωτώ με, δεν θα ήταν καλύτερα να προσπαθήσουμε να έχουμε μια τρίτη ανάγνωση. Διότι εδώ μιλάμε για τον πυρήνα, για το σημαντικότερο στοιχείο της όλης συζήτησης. Ποιο είναι το περιθώριο λιγμού λοιπόν, που μας επιτρέπει το Συμβούλιο για όλα αυτά. Ευχαριστούμε κύριε Ρομεδό. Να σας θυμίσω όμως ότι δεν θα κάνουμε συζήτηση για το θέμα. Απλώς επειδή είχαμε αυτήν την μία ερώτηση, θέλετε κύριε Λούλη να απαντήσετε σύντομα. Ίσως υπάρχει εδώ μια ασφαλμένη ερμηνεία του τι επιδιώκει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο κυρίως επιδιώκει την υλοποίηση της ε, κοινωνικής ασφάλειας που ορίζεται πολύ σωστά στο κείμενο με τρόπο υποχρεωτικό ή εθελούσιο. Δεν λέει ότι δεν θα αποδεχτεί τις εισφορές, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το κείμενο του Συμβουλίου ιδιαίτερος ό,τι αφορά το άρθρο 7, το οποίο εκπροσωπεί ένα στοιχείο προόδου σε σχέση με τα όσα τώρα έχουμε, διότι λέει το κείμενο το Συμβουλίο, όταν υπάρχει σε ένα κάτω μέλος σύστημα κοινωνικής προστασίας για τους αδοτελείς εργαζομένους, για τους ανεξάρτητους εργαζομένους, τα κράτη-μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε διότι εδώ δεν μιλάμε πλέον για συνδύους. Ε, οι ε, συνδύοι λοιπόν, οι σύντροφοι ζωής, θα επωφελούνται της ίδιας κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με το, με το εθνικό δίκαιο. Είναι λοιπόν σαφές, Κοινωνική προστασία προβλέπεται, αλλά μπορεί να γίνει και με τρόπο υποχρεωτικό ή εθελούσιο. για τη δική μας την ε, προτίμηση το καλύτερο ήταν το υποχρεωτικό, αλλά εδώ υπάρχει επιλογή. Είναι σημαντικό και αυτό. Και εξίσου σημαντικό είναι αυτό που λέγεται για την προστασία της μητρότητας. Σε κάθε περίπτωση το κείμενο του Συμβουλίου αποτελεί βήμα προόδου. Σημαντικό μάλιστα σε σχέση με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως σε σχέση με την ισχύουσα οδηγία. Δεν υπάρχει εκεί, δεν γίνεται λόγος για εισφορές και ούτε εδώ τίθεται θέμα εισφορών. Θα διαπραγματευτούμε ακόμη με το Συμβούλιο για να απαλληφθούν κάποια τμήματα κειμένου. Κάποια άρθρα ή εδάφια με τα οποία δεν συμφωνούμε. Και ελπίζω ότι με το Συμβούλιο θα συμφωνήσουμε. Eh, ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστούμε που απαντήσατε στο ερώτημα του κυρίου Ραμέδα. Και ευχαριστούμε που επεξεργαστήκατε αυτό το πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Στη συζήτηση αυτή θα επανέλθουμε τον Απρίλιο και θα ψηφίσουμε στις 4 Μαΐου. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση από την αντιπροσωπεία της Επιτροπής κατόπιν της επίσκεψής τους στην Νέα Υόρκη όπου μιλήσαμε για τη νέα πλατφόρμα της πρωτοβουλίας αυτής ε, Οχτώ μέλη ήταν στην αντιπροσωπεία αυτής που πήγε στη Νέα Υόρκη και τρία επιπλέον μέλη τα οποία ήταν εκεί αλλά δεν ενέπιπταν ε, μέσα στην ποσόστοση. Η διάσκεψη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική όχι μόνο για κοινοβουλευτικά στελέχη αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική για πολλές γυναικείες οργανώσεις παγκοσμίω οι οποίες προετοίμασαν αυτή τη διάσκεψη. Η εναρκτήρια συνεδρίαση έγινε την 1η Μαρτίου, διήρκεσε δύο εβδομάδες και το, η συντονιστική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε στις 4 Μαρτίου θα πιστεύω θα είσαστε ενήμεροι για το ψήφισμα το οποίο υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια. Ξεκινήσαμε με μία συνάντηση πρωινού με την πρόεδρό μας αλλά κάθε μέρα είχαμε και μία συνάντηση follow-up για να ελέγξουμε, να ενημερωθούμε από την Κομισιόν και να ενημερώσουμε την Κομισιόν τι είχε συμβεί εντωμεταξύ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή λοιπόν η ημερήσια ενημέρωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πάρα πολύ σημαντική και ωφέλησε πάρα πολύ την ε, συμβολή τις ε, αντιπροσωπείες μας, τις εργασίες της διάσκεψης. Άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ενδιαφέρει την Επιτροπή μας ε, ήταν ε, μια παράπλευρη δραστηριότητα όπου διάφορες χώρες από διάφορα μέρη του κόσμου είχαν οργανώσει εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, συναντήσεις μαζί με μη κυβερνητικέ οργανώσεις βεβαίως, ε, γυναικείες ε, ενώσεις, ε, γυναικοί σύνδεσμοι και είχαμε τη δυνατότητα λοιπόν να έρθουμε σε επαφή και να ενημερωθούμε μέσω αυτών των παράπλευρων εκδηλώσεων για να ενημερωθούμε για πολλά άλλα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν, μας ενδιαφέρουν. Μετά από την επίσκεψη αυτή της αντιπροσωπείας, εγώ ως επικεφαλής αντιπροσωπείας είχα την ε, δυνατότητα να συμμετάσχω ως παρατηρητής ε, κατά τη διάρκεια των εργασιών. Και νομίζω ότι για την Επιτροπή μας ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία. Μας δόθηκε η δυνατότητα ε, να συμμετάσχουμε στις εργασίες ως παρατηρητές και έτσι μπορέσαμε να ενημερωθούμε να, για τις εργασίες, να δούμε πώς εξελίχθηκαν, τι ελέγχθη, τι ήταν η ημερήσια διάταξη. Θα σας ενημερώσω τώρα σε τι ε, συνεδριάσεις, σε τι συναντήσεις ε, συμμετέσχαμε ε, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. συναντήσαμε την κυρία Σάλι Βέγγεν Βάιτς, η οποία είναι διευθύντρια της αναπτυξιακής ομάδας ε, του ΟΗΕ. Επίσης την κυρία Ρέιτσελ Μαριάνια, η οποία είναι αναπληρώτρια, γραμματέας και ειδική σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θέματα, σε θέματα οικολογίας, οικολογικά και συζητήσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση, δηλαδή αν θα πρέπει ο ΙΕ να δημιουργήσει... Α, η, η, η, η κυρία ήταν ειδική σύμβουλη σε θέματα ισότητος ισότητος. Και αν θα πρέπει, συζητήσαμε ο ΙΕ να δημιουργήσει ένα δίκτυο, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συζητούνται όλα τα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων. Υπήρχε λοιπόν ένα μεγάλο ενδιαφέρον και πλούσιο πρόγραμμα παράπλευρων συνεδριάσεων παράλληλα με τις εργασίες ε, της, της διάσκεψης και έχετε βεβαίως ε, την ε, έκθεση, μια συνοπτική έκθεση της επίσκεψής μας, της επίσκεψη και τη συμμετοχής της αντιπροσωπείας μας, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε πλήρως. Απλώς ήθελα τώρα να ρωτήσω εάν ε, στα πλαίσια της πλατφόρμας του Πεκίνου και του Beijing συν 15 υπάρχει καμία ερώτηση ή σχόλιο. Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα. Ε, το τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως Επιτροπή. Πρώτον, πρέπει να συζητήσουμε, τις, ε, τις, να συζητήσουμε το, τα θέματα που συζητήθηκαν μέσα στον ΟΗΕ με την κυρία Ρέτσελ Βάιτ για την ε, διάσταση του φύλου. Έχει δημιουργηθεί μια πολύ περίεργη κατάσταση όπου έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το πλαίσιο της διάστασης του φύλου και όλες οι εργασίες έχουν συγκεντρωθεί στα χέρια ενός οργανισμού και δει στα πλαίσια της UNIFEM. Ε, λοιπόν, πιστεύω ότι ορισμένες χώρες κρατώνται σε ομοιρία, διότι ένας φορέας λαμβάνει τις αποφάσεις, οι υπόλοιπες χώρες είναι όμοιροι των αποφάσεων αυτών και δεν υπάρχει ισότιμη συμμετοχή. Μας ζήτησαν λοιπόν να σήξουμε αυτά τα θέματα σε διάφορες αντιπροσωπείες. Από όλα τα μέρη του κόσμου, παραδείγματος χάρη με τις χώρες της ε, Νότιας Αμερικής, με αφρικανικές χώρες για να ε, μπορέσουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε αυτήν την περίεργη κατάσταση. Το θέμα άπτεται βεβαίως των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ. Είχα την εντύπωση ότι πολλοί συμμερίζονται αυτή την άποψη, ότι δηλαδή ε, έχει φτάσει πλέον, έχει οριμάσει ο χρόνος να λύσουμε ή να συζητήσουμε από εδώ και πέρα τα θέματα πολυμερός και όχι μόνο μονομερός, συγκεντρωμένα δηλαδή σε έναν οργανισμό. Δεδομένου δε ότι ήμασταν, είχαμε το καθεστώς του παρατηρητή, πιστεύω ότι η κυρία Επίτροπος Άστον θα πρέπει να ασκήσει πίεση για να μπορέσει να ακούγεται σωστά η φωνή μας και έντονα με τις απόψεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάρτερ Μπάουερ για τις απόψεις σας. Υπάρχουν άλλα μέλη τα οποία θα ήθελα να σχολιάσουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της αντιπροσωπείας μας που πήγαν και συμμετείχαν στην επίσκεψη αυτή στη συνάντηση της πλατφόρμας, διότι επιτελούμε σημαντικό έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ακόμη πολλά από που μένουν να γίνουν, όμως είναι πραγματικά σημαντικό να συμμετέχουμε σε αυτό το παγκόσμιο κίνημα. Από τα λόγια σας, σημειώνω αυτά που μας είπατε, όπως και η Edith Bauer, πρέπει να αναλάβουμε την πραγματική αυτή ευθύνη που μας αναλογεί. Και από από το γεγονός ότι ο ΙΕ προβλέπει μία δομή που εργάζεται και για την ισότητα των δύο φύλων, εκεί μπορούμε να διαδούμε ένα σημαντικό βήμα. Δημιουργούνται σιγά σιγά διάφοροι κρίκοι τη αλυσίδας, της φάσης μιας διαδικασίας. Θα χρειαστεί λοιπόν να είναι ενεργή η αντιπροσωπεία μας, τα μέλη της δηλαδή, και να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις ε, πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να τονίσω ότι πράγματι είναι σημαντικό να έχουμε όλους αυτούς τους κρίκους της αλυσίδας, ώστε να είναι αυτή η αλυσίδα γερή. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουν όλα τα μέλη της Επιτροπής μας, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό το ζήτημα εφ' εξής. Ε, με πολλές ευχαριστίες λοιπόν σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν την επίσκεψη και στη γραμματεία που με το τεράστιο έργο της φρόντισαν να έλθουν πέρα σε όλα τα διοργανωτικά της επίσκεψης αυτής και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το ταξίδι αυτό ήταν μια σοβαρή κίνηση γιατί με την συμμετοχή μας στις διάφορες συναντήσεις μπόρεσαν ε, τα μέλη ενεργά να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης, το υπαριθμόν 5, όπου έχουμε τις βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει. Εφαρμογή του Προγράμματος Εργασίας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010. η πορεία του θέματος αυτού και ο λόγος που το προβλέψαμε στην ημερήσια διάταξη είναι ότι οι συντονιστέ αποφάσισαν τον Ιανουάριο αποφάσισαν τον Ιανουάριο να αποφάσισαν από κοινού με τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού να υποβληθούν τροπολογίες για την γνωμοδότηση αυτή στην Επιτροπή πολιτισμού που είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό μαζί με την ε, δική μας την Επιτροπή. Η κυρία Χάνιμπαλ ε, υπέβαλε έξι τροπολογίες και εφόσον είναι μαζί μας η συνάδελφος θα μας μιλήσει για αυτές τις έξι τροπολογίες της. Ο στόχος αυτής της συζήτησης σήμερα είναι να ψηφίσουμε για αυτές τις έξι τροπολογίες εφόσον όλοι συμφωνήσουμε και αν εγκριθούν οι τροπολογίες αυτές θα ψηφιστούν και στην Επιτροπή Πολιτισμού. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Χάνιμπολ στον συνεδρίασή μας και τη δίνω Γεια σας. Καλό απόγευμα. Ζητώ συγγνώμη που άργησα. Θέλω λίγα λεπτά να σας παρουσιάσω τις τροπολογίες. Όπως ξέρετε αυτή η έκθεση αναθεωρεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2010 και τα συγκριτικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αναθεωρηθεί από τότε. Πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε, να τα κοιτάξουμε και να τα επικαιροποιήσουμε, να δούμε ε, επίσης αν έχει επιτευχθεί πρόοδος και γι' αυτό έχω παρουσιάσει αυτές τις ε, τροπολογίες. Όπως ξέρετε είμαι μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού, είμαι και συντονίστρια της Επιτροπής Πολιτισμού Είμαι επίση το μέλο από την Επιτροπή Πολιτισμού που είναι υπεύθυνο για τη διάσταση του φίλου. Γι' αυτό ακριβώς παρουσίασα αυτές τις έξι τροπολογίε. Ο στόχος μου είναι να ενισχύσω, να τονίσω αυτά τα οποία ήδη έχουμε συζητήσει και ζητήσει. Και να αυξήσουμε το ποσοστό ανδρών ή γυναικών εκεί όπου υποεκπροσωπούνται και ε, δεδομένου ότι όπως όλοι ξέρουμε οι γυναίκες αμείβονται στα περισσότερα επαγγέλματα λιγότερο να βελτιώσουμε την κατάσταση και που υπάρχει ανισορροπία στη διάσταση του φύλου μέσα στα πλαίσια και της κοινωνικής συνοχής. Πρέπει λοιπόν να ενταχθούν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας και να εξασφαλίσουμε ότι ορισμένοι τομεί εργασίας δεν αποκλείουν τις γυναίκες. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Χάνιβαλ. Νομίζω ότι ο... η πρόταση αυτή είναι καλή, έτσι όπως παρουσιάζεται, και ότι μας διευκολύνει την παρουσία μας ε, και το, τη, τη, φωνή μας, το άκουσμα της φωνής μας και σε άλλες, υπηρεσίες, σε άλλες επιτροπές. Συγγνώμη. Δεν ε, νομίζω να επισημεί κανείς να σχολιάσει αυτή την πολύ σύντομη παρουσίαση, άρα πιστεύω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα αυτές τις τροπολογίες της κυρίας Hannibal. Παράγραφος 4α λοιπόν, υπέρ, Ψηφίζουμε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Ε, εγκρίθηκε. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Ε, ε τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν κυρία Χάνιμπολ και Υιοθετήσαμε τώρα τις τροπολογίες αυτές, οι οποίες θα υποβληθούν στην Επιτροπή Πολιτισμού. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το θέμα 6. Πτυχές σχετικές με την ισότητα των φύλων στην περίοδο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ε, αποφασίστηκε να συζητηθεί το θέμα αυτό από την Επιτροπή μας και έχουμε ε, την, τον κύριο Ρομέμπα που είναι υπεύθυνο για αυτό το θέμα και πιστεύω να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σήμερα επί του θέματος. Εν συνεχεία, βάση του χρονοδιαγράμματος στις 23 Μαρτίου είναι η προθεσμή υποβολής τροπολογιών και το 24 Μαΐου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή και ελπίζω να παρουσιαστεί στην Ολομέλεια τον Ιούλιο για προσψήφιση. Θα ήθελα να ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, το, τον εισηγητή μας και τι έχει να πει επί του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το θέμα αξίζει να συζητηθεί και ίσως θα πρέπει και να γίνει αυτή η δουλειά πιο νωρίς γιατί κάποια στιγμή δεν συζητούμε πώς να αποφύγουμε την κρίση αλλά πώς θα βρούμε διέξοδο. Οπότε Γι' αυτό ακριβώς και μας χρειάζεται να μπορέσουμε να δούμε τα πράγματα και από το πρίσμα αυτό της ισότητας των φίλων, Να δούμε τι ευθύνες υπάρχουν σε σχέση με τις συνέπειες της κρίσης και επίσης να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, τι επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν τόσο ώστε να βρούμε έξοδο στο αδιέξοδο αυτό. Επομένω να κάνουμε να δούμε και αυτήν την τη γωνία. Θα πρέπει όμως να άρουμε αυτό το κενό το οποίο υπάρχει, κενό στην ανάλυση, αλλά και αυτό που λείπει και από τις σχετικές προτάσεις. Αν κάτσει κανείς και δει τους τελευταίους μήνες τι γράφει ο τύπος για την ε, κρίση, αυτό το οποίο αναδεικνύονται είναι τα εξή. Πρώτα-πρώτα, χτύπησε αυτή η κρίση βασικά κάποιους κλάδους. Λέω, επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μερίδα του τύπου. Επαναλαμβάνουμε επομένω ότι κυρίως αυτή η κρίση χτύπησε κάποιους κλάδους της οικονομίας καταρχήν ε, που κυριαρχούνται από τους ε, άντρες σε σχέση με αυτό, με την, την, την, ε, την, την κρίση, γιατί από την άλλη μεριά έχουμε εδώ πέρα και αυτό το ότι θα πρέπει να συρρυκνωθεί η δαπάνη του δημοσίου και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε ότι οι γυναίκες είναι επίσης ευάλωτη θέση στις περισσότερες αν όχι όλες τις χώρες. Να μια πρώτη σκέψη. Αν κάτσουμε και να λύσουμε αυτά τα θέματα τότε θα καταλάβουμε ότι πρώτο πρώτο. Λείπει μια ανάλυση του πώς η κρίση χτυπάει όχι εκείνους τους κλάδους που αναφέρθηκαν συγκεκριμένες βιομηχανίες την αυτοκινητοβιομηχανία Φερρυπίν ή σε κάποιες χώρες ας πούμε όπως την Ισπανία τον κατασκευαστικό οικοδομικό τομέα που είναι όλοι αυτοί οι κλάδοι που κυρίως απασχολούν άντρες. Όμως αυτό το οποίο λείπει ότι κανεί δεν έχει κάτι να δει τι γίνεται στου κλάδου όπου υπάρχουν γυναίκε εργαζόμενε. Εκεί είναι πάρα πολύ προσωρινά εργαζόμενοι γιατί είναι κάποιες δραστηριότητες σε αυτούς τους κλάδους που η δουλειά γίνεται κυρίως από γυναίκες. Στη δε αλυσίδα, αλληλουχία των συνεπειών της κρίσης κάποια στιγμή θίγεται και η γυναίκα και όχι μόνο ο άντρας. Θυμάμαι ότι είχαμε πάει στην ε, χώρα των Βάσκων πριν από λίγες μέρες με την Επιτροπή ελίας και εκεί συναντηθήκαμε με διάφορους εκπρόσωπους του κλάδου αυτού των Θεσσαλίας. Ε, οπότε συζητήσαμε τα προβλήματα και τις λύσεις. Επίσης ε, κάτσαμε και συνθήκαμε και κάποιες ε, γυναίκες και τις εκπροσώπους τους που ασχολούνται με το, με, με το ράψιμο των δικτυών τα οποία σκίζονται. Αντίχεια δηλαδή του ψαρέματος. Δύσκολη δουλειά σε δύσκολες συνθήκες. Όμως θα πρέπει να δούμε ότι σε τέτοια δύσκολη συγκαιρία από κάποιο μετασχηματισμό αξίζει να αναγνωριστεί η δουλειά αυτή που είναι τόσο απαραίτητη για την αλληλευτική δραστηριότητα γιατί χωρίς αυτές τις εργαζόμενες δεν θα μπορούσε να βγει να ψαρέψει ο ψαράς. Να ένα παράδειγμα επομένως το πώς δεν προβάλλεται, δεν φαίνεται ο ρόλος, η δουλειά της γυναίκας και το σούτο μάλλον στην εποχή κρίσης που οι επιπτώσεις είναι πιο έμεσες χτυπιούνται πρώτα κάποιοι άλλοι κλάδοι, δηλαδή, όμως στη συνέχεια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οπότε και αντίστοιχα, εάν δεν προβάλλεται ο ρόλος σου, είναι ακόμη πιο δύσκολο να, να βρεις μια λύση από ότι κάποιος που πιο άμεσα θίγεται και πιο άμεσα φαίνεται. Θα πρέπει εμένα να προβληθούν μια τέτοιε δραστηριότητε. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε αυτού του κλάδου δραστηριότητα. Ε, αυτά τα οποία αναδεικνύονται ε, από την συζήτηση του προβληματισμού για την κρίση, αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν ε, αναγνωρίζονται και αυτά να καλυφθούν, αυτές, αυτά τα προβλήματα να καλυφθούν από όποιε λύσει ανεβρίσκονται ή προτείνονται. Είπαμε ότι η κρίση ξεκίνησε από τον χρηματοοικονομικό τομέα. Οπότε βλέπουμε όμως ότι πάλι και η χρηματοδότηση από εκεί θα, θα προέλθει και φυσικά μιλάμε για κάποιο τομέα που κυριαρχείται από τους άντρες σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι βασικές τράπεζες, η ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ταμείο ε, έχουν επικεφαλής άντρες. Όμως, όσον αφορά τα διοικητικά συμβούλια αυτών των βασικών μεγάλων τραπεζών έχουμε 16% των μελών των διοικητικών συμβουλίων που είναι γυναίκες. Βλέπουμε επομένω πρώτο στοιχείο ανισότητας όσον αφορά τα της διοίκησης αυτών των βασικών τραπεζών. Για να δούμε πιο πολύ εις βάθος. Lehman Brothers και όχι Lehman Sisters λεγόταν, ε, γιατί μου επιτρέψει ένα φτηνό αστείο. Θα ήταν όμως η ίδια η κρίση αν λεγόταν Lehman Sisters. Μπορεί κανείς να κάνει μια διαφορετικές ε, αναλύσεις ανάλογα με τις ε, πεπιθήσεις του και τις απόψεις του. Όμως θα διαπιστωθεί ότι στις τράπεζες που υπάρχει περισσότερο όταν δύο φίλων, εκεί, εκεί χτυπήθηκε λιγότερο εργαζόμενος από την κρίση από σε, σε κάποιους οργανισμούς τραπεζικούς όπου υπήρχε ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επομένως θα πρέπει να ληφθούν κάποια δραστικά μέτρα όσον αφορά κάτι που το έχουμε αναλάβει επανειλημμένα. Αλλά και εδώ έχει σχέση με το πώς θα υπάρχει περισσότερη ισότητα στις ε, ρυθμιστικές αρχές, οι διαχειριστικές αρχές, εκεί που υπάρχει η πιο βασική πολιτική ή οικονομική εξουσία. Και έχουμε κάποια παραδείγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, τα λέμε στην έκθεση, ας πούμε στην Ισλανδία. Στην Ισλανδία, εκεί αξιοποιήθηκε πάρα πολύ μια τέτοια πρωτοβουλία για την ισότητα, ούτω ώστε να αρθεί η ανισότητα για τη λήψη αποφάσεων. Και στη Νορβηγία 40% αποφασίστηκε να είναι συμμετοχή των γυναικών στα όργανα διοίκησης. Να κάτσουμε να δούμε επομένω τι ευθύνε υπάρχουν και να διορθώσουμε την κατάσταση. με τη χρηματοπιστωτική κρίση. Τελευταία σκέψη τώρα είναι η εξή. Όσον αφορά τις διορθωτικές κινήσεις που γίνονται σε ορισμένε περιπτώσεις, αλλού δε ε, έχουμε κάποιες επενδύσεις που οδηγούν στην έξοδο από την κρίση, να δούμε πώς θα έχουμε ένα καινούργιο πλαίσιο κοινωνικό-οικονομικό και κατά αυτόν τον τρόπο να βάλουμε τι βάσει για ένα καινούργιο οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο. Πρώτη σκέψη. Όταν μιλούμε για αυτές τις θέσεις στην αγορά ή τις ευκαιρίες στην αγορά και μας οδηγούν στην δημιουργία θέσεων εργασίας που είναι πάρα πολύ βασικό και για μας είναι σε συνέχεια του New Green Deal, οι πράσινες θέσεις απασχόλησης, που έχουν άμεση σχέση με την καθαρή ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την μείωση των εκπομπών του διοξιδίου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι εάν αυτές οι ενέργειες δεν γίνουν συμπληρωματικά με προώθηση περισσότερης παρουσίας συμμετοχής γυναικών, περισσότερης ισότητας, εάν δεν γίνουν όλα αυτά, τότε θα επαναλάβουμε τα λάθη τα οποία έγιναν στο παρελθόν και μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση. Άρα, δημόσιες επενδύσεις εκεί που έχουμε αυξημένη συμμετοχή ανδρών. Αλλιώς έχουμε επανάληψη και όχι διόρθωση των λαθών του παρελθόντος. έτσι. Έχοντας υπόψη την επιδιωκόμενη ισότητα. Υπάρχει κάτι άλλο όμως, το οποίο πολλές φορές το ξεχνούμε, είναι ότι σε κάποιους τομείς όπου έχουμε ευξημένη συμμετοχή των γυναικών θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η συμμετοχή των γυναικών. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε ακούσει σχετικές προτάσεις ακόμα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ενώ κυρίως την ε, Επιτροπή, αλλά ούτε από το Συμβούλιο. Και έτσι να αξιοποιήσουμε αυτές τις, αυτούς τους κλάδους, αυτές τις δραστηριότητες που κυρίως του κρατικού τομέα όπου θα πρέπει να επενδύσουμε την κοινωνική υποδομή. Έτσι θα έχουμε νέες ευκαιρίες για να μπορέσουμε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, να διορθώσουμε τις ανισότητες και αποκλήσεις της αγοράς απασχόλησης. Μας δίνεται αυτή η ευκαιρία για να προχωρήσουμε από πλευράς ισότητας των δύο φύλων. Μέσα από αυτή την προβληματική που αναπτύσσεται εδώ στο Κοινοβούλιο, ισότητα ευκαιριών, ισότητα των δύο φίλων, μέσα από την έκθεση αυτή. Να κατεβάσουμε κάποιες προτάσεις, να δώσουμε κάποιες ιδέες και έτσι να δούμε πώς θα διορθώσουμε κάποια λάθη διαρθρωτικά και έτσι θα βγούμε από την κρίση. Αλλιώς θα πληγούμε ακόμη περισσότερο από τις αρνητικές συνήπεις της κρίσης που χτύπησε πολύ περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες. Άλλωστε, όλο ένα και περισσότερο αυξάνει η παρουσία της γυναίκας στην ε, αγορά εργασίας. Εκτός από την αυξημένη παρουσία τους όμως, είναι και πιο ευάλωτες οι γυναίκες. Περισσότεροι ανασφάλεια έχουν και εργασιακή και από πλευρά των συμβάσεων εργασίας που έχουν και απλώς νομική επομένω Πρέπει να συγκεράσουν την ε, οικογένεια με τη δουλειά. Οπότε θα πρέπει αυτό το ζήτημα να ειδωθεί και στα πλαίσια του ορίζοντα του 2020. Εδώ μπορεί να αναδειχθεί ο ρόλος της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ούτω ώστε και το πρόβλημα να εξαστεί από αυτή την οπτική γωνία, αλλά και να επιζητηθούν έτσι οι λύσει. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Δεν έχουμε ομιλητές. Εγώ όμως είμαι σκιώδης εισηγήτρια από την πλευρά των σοσιαλιστών και δημοκρατών, δημοκρατών και σοσιαλιστών, οπότε θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας αφορά ένα ζήτημα σοβαρότατο και μεγάλης ε, επικαιρότητα. Όπως υπόθηκε από τον εισαγητή, αυτή η κρίση κυρίως προκλήθηκε από άνδρες. Αναφερθήκατε στην ε, ισχνή παρουσία των ε, γυναικών στα τρία βασικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τραπεζικούς δηλαδή οργανισμούς, αλλά αυτή η ελλειπής ε, αντιπροσώπευση ε, είναι κάτι που εκδηλώνεται και σε εθνικό επίπεδο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ε, κρατών μελών. Αρκεί να πούμε ότι καμία από τις κεντρικές τράπεζες των 27 κρατών μελών δεν έχει πρόεδρό της γυναίκα. Σε όλες τις περιπτώσεις πρόεδροι είναι άντρες. Επίσης αληθεύει ότι οι γυναίκες πλήττονται κατά κύριο λόγο εκείνες. Είναι τα βασικά θύματα της κρίσης. Αυτή τη στιγμή και περισσότερο εργάζονται προσωρινά και λιγότερο καλύπτονται από τα συστήματα της κοινωνικής ασφάλειας. Και μιλήσατε κι εσείς για το ευάλωτο της εργασίας τους, επίσης για την ελληπή συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων τόσο οικονομικών όσο και διοικητικών. Επίσης, ε, στην απασχόληση ανδρών και γυναικών αυξήθηκε η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Από το 15% φτάσαμε στο 16,2% στον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο. Κατά τα άλλα, σημαντικό είναι να συλλογιστούμε, να σκεφτούμε, να διαδούμε λύσεις για το πώς μπορούν οι γυναίκες να βγουν από αυτήν την κρίση. Ποια είναι η διέξοδος, δηλαδή να υπάρχει μια διπλή προοπτική. Από τη μια να έχουμε κατά νου ότι η κρίση πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και από την άλλη θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να στηρίξουμε ιδίως τις γυναίκες για να βγουν από την κρίση. Στην συνεισφορά των γυναικών για την διέξοδο από την κρίση καλό είναι να έχουμε υπόψη και κάποιες μελέτες που έχουν εκπονηθεί. μελέτες που καταδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερο αριθμό γυναικών στο διοικητικό τους συμβούλιο έχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερες επιδόσεις στο χρηματιστήριο αξιών όσες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά και ως προς το κέρδος, δηλαδή τα αποτελέσματα των πωλήσεων μεταξύ 70 έως 80% προστιθε... 85% μάλλον προστιθέμενη αξία. Διαφορά δηλαδή, καλύτερα αποτελέσματα. <clears throat> και μιλάμε για επιχειρήσεις αξιόπιστες που έχουν ε, τέτοια αποτελέσματα, όπως η μελέτη που ετοίμασε η Catalyst και αποδεικνύει κάτι τέτοιο, μια αρκετά αξιόπιστη εταιρεία μελετών. Έπειτα, τον επενδύει στις γυναίκες ως εργαζόμενες είναι και πιο αποδοτικό αλλά όχι μόνο για την επιχείρηση, για την κοινωνία γενικότερα. Διότι οι γυναίκες οι ίδιες επενδύουν περισσότερο στην ε, σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους, άρα βελτιώνουν την λήψη προσόντων των παιδιών, την ε, ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, την επαγγελματική τους μελλοντική σταδιοδρομία και έτσι έχουν και σοβαρή συμμετοχή στην διαχείριση του προπολογισμού, του οικογενειακού προπολογισμού. Μια τελευταία παρατήρηση από πλευρά μου είναι ότι πέραν των όσων ήδη είπαμε και των παραδειγμάτων ε, της Νορβηγίας λόγω χάρη, αλλά και της Γαλλίας, όπου Στη Γαλλία βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία ποσόστοσης 40% να αποδοθεί στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, των κρατικών και των εισηγμένων στο χρηματιστήριο στις γυναίκες. Οπότε δεν είναι μόνο το σύστημα των ποσοστώσεων ε, στην δεν μπορεί να βρει μάλλον το σύστημα των ποσοστώσεων ε, εφαρμογή μόνο στο πολιτικό βίο, αλλά μπορεί να βρει και στην οικονομική σφαίρα εφαρμογή. Επίσης να πω ότι σε ό,τι αφορά την στρατηγική του 2020, όπου ήδη διαβλέπουμε νέους δρόμους, ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό το νέο μοντέλο, το νέο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την συμμετοχή των γυναικών από τη μια, αλλά και τις συνέπειες των νέων οικονομικών πολιτεών, πολιτικών που σχεδιάζονται. Γνωρίζουμε ότι καμία πολιτική δεν μπορεί να έχει τον ίδιο αντίκτυπο στις γυναίκες και στους άντρες με τον ίδιο τρόπο. Οι επιπτώσεις είναι πάντα διαφορετικές ανάλογα με το φύλλο. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη και να ληφθεί σοβαρά υπόψη και στην χάραξη της πολιτικής του 2020. Το νέο αυτό πρότυπο θα πρέπει λοιπόν να καλύπτει και την συμμετοχή των γυναικών, το ρόλο τους στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους κρατών μελών και όλου του κόσμου. Ήδη τώρα έχουμε και άλλους ομιλητές και τώρα η κυρία Μωρά Σαρτιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπόθηκαν ε, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για αυτή την ε, έκθεση και πολλά ενδιαφέροντα περιέχει κιόλα. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρωμέβα λοιπόν και την κυρία Εστρέλα για τις συμπληρωματικέ της παρατηρήσεις, γιατί πολλά από τα σοβαρότερα ζητήματα έχουν ήδη καλυφθεί. Ιδιαιτέρως, όπως και εσείς είπατε κυρία Εστρέλα, μόλις τώρα, το θέμα της απουσίας, της πλήρους απουσίας των γυναικών από σοβαρές ε, θέσεις ευθύνη τόσο στο ευρωπαϊκό επίπεδο και το διεθνές, αλλά και στο εθνικό, τον καθενός από τα κράτη-μέλη μας. Μιλήσατε για τις ε, μισθοδοτικές διαφορές και αναφέρατε ποσοστά. Αυτό θα πρέπει να το δούμε με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία στη διάρκεια ενός έτους. Γιατί για να κερδίσει μια γυναίκα τον ίδιο μισθό με έναν άντρα από την 1η Ιανουαρίου στον 31η Δεκεμβρίου, η ίδια γυναίκα θα πρέπει να δουλέψει ως τις 26 Μαρτίου της ερχόμενης χρονιάς. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, Πρόεδρε? Σημαίνει ένα τρίμηνο παραπάνω ετησίως. Παρά τέσσερις μέρες, τέλο πάντων. Αλλά είναι ένα τρίμηνο ετησίως. Φανταστείτε την μισθοδοτική διαφορά και την ε, ζημία την οικονομική αυτή κατά των γυναικών και προς όφελος των ανδρών. Δεν θέλω εδώ να είμαι φεμινίστρια στην προσέγγιση μου, αλλά βλέπω τα πράγματα από την άποψη της ισότητας, της δικαιοσύνης μεταξύ πολιτών. Οι ίσες ευκαιρίες, η ίση εργασία σημαίνει και ίσο μισθό. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η σημερινή κρίση που πλήττει περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρες όπως το αποδείξατε, να γίνει μια ευκαιρία ώστε να αναλάβουμε κι εμείς πολύ περισσότερες πρωτοβουλίε, ενέργειες, ώστε η μισθοδοτική αυτή απόσταση να μειωθεί. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να επιληθούν αυτά τα θέματα και να έχουμε πολύ σαφείς στόχους. Ζητήσατε, και ήδη αυτό εν μέρη προβλέπετε, αλλά πρέπει οπωσδήποτε με τρόπο εμπεριστατωμένο, με στατιστικά στοιχεία για άντρε και γυναίκε, να το στηρίξουμε. Γι' αυτό εργαζόμαστε, αλλά πρέπει να πάμε ακόμη παραπέρα. Ιδίω στην κάλυψη τη μισθοδοτική αυτή απόσταση. Οι γυναίκε δεν μπορεί πλέον να το δέχονται αυτό. Δεν μπορεί να δέχονται τέτοια μεταχείριση στο επίπεδο τη μισθοδοσία. Και επιπλέον, και για μένα αυτό είναι το θεμελιώδε στοιχείο που δυστυχώ δεν το βρίσκω στην έκθεσή σα, κύριε Ρωμέδα, και θα ήθελα να το περιλάβετε. Είναι το εξή, ότι το, το πρόβλημα ουσιαστικά είναι ότι οι γυναίκες έχουν και περισσότερα πτυχία συνήθως από τους άνδρες. Θα σας το αποδείξουν αυτό όλες οι στατιστικές. Συνεργαστήκαμε με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και εκπονήσαμε μελέτη για το θέμα αυτό και με άλλες δομές οι γυναίκες έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Peut-on expliquer ce que je viens d'entendre? Que dans la crise Πώ είναι δυνατόν αυτά τα δύο να συμβιβάζονται. Κατά τη διάρκεια τη κρίση, οι γυναίκε να έχουν ε, εργασίε μερική απασχόληση, να ε, να υπομισθώνουν τη θέση εργασία του και από νομική άποψη να μην καλύπτονται. Αυτό το σημείο θέλω να αναφέρετε στην έκθεσή σα, κύριε Ρωμέβα. Διότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο αυτό το πρόβλημα. Η κρίση ήταν ε, μια ισχυρή ένα ισχυρό κλονισμό για να αναγκαστούμε να δούμε τη ρίζα του προβλήματος. Εάν δεν το κάνουμε τώρα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020, τότε ας πούμε ότι ερχόμαστε στις συνεδριάσεις για την ευχαριστησή μας, για τη διασκέδασή μας και ότι δεν θα κάνουμε τίποτα επί της ουσίας. Το πρόβλημα αυτό της αναλογίας μεταξύ μερφωτικού επίπεδου και επίπεδου απασχόλησης εργασιακής ε, αποκατάστασης είναι κάτι που πρέπει να το συμπεριλάβουμε στη συζήτηση. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να προσεγγίσουμε και ένα δεύτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτού που, της καταπολέμησης αυτού που ονομάζουμε γυάλινη οροφή. Ένα είδος ε, περιορισμού Τόσο στην κοινωνία, <clears throat> εδώ δεν με ενδιαφέρει να επιρρύψω ευθύνε όσο να εξεύρουμε λύσει, ένα λοιπόν είδο περιορισμένο φραγμού στην κοινωνία που δεν επιτρέπει στι γυναίκε να προοδεύσουν. Είτε στην ιδιωτικό τομέα, είτε στο κρατικό μηχανισμό. Νομίζω λοιπόν ότι το, να καταπολεμήσουμε την γυάλινη οροφή στην εκπαίδευση, στην διαβίου κατάρτιση, διότι αν αρχίσουμε να κοιτάζουμε μόνο την εκπαίδευση, θα πρέπει να σκεφτούμε τα αποτελέσματα, θα τα δούμε στα εγγόνια μας. Να είμαστε λοιπόν πιο δραστήριοι στην ε, στρατηγική 2020 και να σκεφτούμε ότι η διαβίου κατάρτιση θα είναι μια ευκαιρία ώστε οι γυναίκες να απελευθερωθούν, να μπορέσουν να πάνε ακόμη παραπέρα. Το αποδεικνύουν και τα στατιστικά στοιχεία. Είναι λοιπόν σοβαρό το ζήτημα. Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να καλύπτεται στην έκθεση και δεν βρίσκω να παρουσιάζεται όπως εγώ θα το ήθελα, είναι ότι το παράδειγμα θα πρέπει να το δίνει ο δημόσιος τομέας. Η κυρία Στρέλα είπε ότι στη Γαλλία θα υπάρξουν ποσοστώσεις και για τις επιχειρήσεις, του 40%. Σαφώς, Ωραία είναι η ιδέα. Όμως γιατί να πάμε να ζητάμε από τους ξένους να κάνουν κάτι που δεν κάνουμε εμείς. Γιατί ο δημόσιο τομέας να ζητάει από τον ιδιωτικό να κάνει κάτι που ίδιος δεν το πράττει. Υπάρχουν πολλές γυναίκες και στον κρατικό μηχανισμό. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτόν τον τομέα και όταν α, δει ε, τα κλιμάκια, όταν μάλλον ανέβει κανείς τα κλιμάκια, βλέπει ότι οι γυναίκες δεν εμφανίζονται. Όσο πιο ψηλά πάει κανείς στην ιεραρχία ο δημόσιο λοιπόν τομέα να δίνει το παράδειγμα. Αυτή είναι τρίτη μου επιθυμία και θα ήθελα και πάλι και στη στρατηγική 2020 να υπάρξει και αυτό ο στόχο. Η τέταρτη παρατήρησή μου είναι μία παραδοχή για τις ποσοστώσεις. Πρέπει να παραδεχτώ ότι όταν προέβλεψε τις ποσοστώσεις η Γαλλία στον πολιτικό βίο, εγώ ήμουν αρκετά επιφυλακτική. Διότι οι ποσοστώσεις, αν θέλετε, σημαίνουν ότι υπάρχει ένα, ένα όριο προστασίας για κατηγορίες που όμως φαίνονται έτσι και εμφανίζονται αδύναμες. Εγώ νομίζω ότι εφόσον υπάρχουν ίσες αρμοδιότητες και ικανότητες, πρέπει να υπάρχουν και ίσες ισότιμες θέσεις. Θα είναι περίπου καμιά δεκαετία που ελήφθησαν αυτά τα μέτρα. Τώρα με τη χρονική απόσταση πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι οι ποσοστώσεις τελικά βοηθούν. Βοηθούν να επιτύχουμε περισσότερο, περισσότερη ισότητα. Δεν λέω ότι αυτό αρκεί, δεν λέω ότι πρέπει να παραμείνουμε στη μέθοδο των ποσοστώσεων. Ακούω πολλά παράπονα από την πραγματικότητα οι πολλούς που λένε ότι οι γυναίκες ναι, μπορεί να μην είναι αρκετά ικανές αλλά τις βάζουμε νούμερο 2, νούμερο 4 αυτό με στενοχωρεί διότι εγώ βλέπω πολλές γυναίκες ικανότατες γυναίκες ικανότατες που απελευθερώνονται για να λάβουν τη θέση που τους αξίζει αλλά δεν είναι πολλέ. Δεν είναι πολλέ. και νομίζω ότι οι ποσοστώσει από, από μόνες τους δεν αρκούν. Στην πραγματική πολιτική μαζί με άλλους μοχλούς. Όπως αυτούς που βλέπω και αυτού που σας ζήτησα, ναι τότε μπορεί να είναι ένας τρόπος να πάμε προς το στόχο. Αλλά όχι αυτός σκοπό. Και τέλος, κάτι για το οποίο θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, είναι ο συνδυασμό του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο. Εδώ στου στόχου τη στρατηγικής του 2020 να μην ξεχνάμε ότι του πραγματικού μοχλού θα τους ορίσουμε εμεί ως στοιχεία για την συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πλόμ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία που επιτέλεσε. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά καλά σημεία, πολλές ουσιαστικές παρατηρήσεις και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο ανέλευε μια τέτοια έκθεση ιδίες πρωτοβουλίες. Υποστηρίζω πλήρως τον, τη συνάδελφό μου κυρία Στρέλα αλλά και την κυρία Σαρτιέ. Θα ήθελα μόνο να παρατηρήσω ότι βέβαια το θέμα των ίσων ευκαιριών είναι, θα πρέπει να αποτελέσει ένα σαφέστατα καθορισμένο και οριοθετημένο κεφάλαιο για το μέλλον. Και πολλές φορές το θέμα αυτό κυριολεκτικά καίει τις γυναίκες, ιδιαίτερα όσον αφορά την πτυχή της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Συμφωνώ επίσης ότι ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα στο θέμα της ισότητας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στη Ρουμανία αυτή τη στιγμή προβλέπεται η απώλεια πολλών θέσεων εργασίας και αυτές οι θέσεις εργασίας θα κοπούν κυρίως εκεί που δουλεύουν γυναίκες. 15.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν αυτό το μήνα και το 85% αυτού του αριθμού θα θα είναι θέσεις τις οποίες καλύπτουν γυναίκες. Πολύ ψηλό ποσοστό λοιπόν απώλειας θέσεων εργασίας για τις γυναίκες. Αυτό ήθελα να το πω για να εστιάσουμε την προσοχή μας. Ε, ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Όταν γίνονται περικοπές θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα, το πρώτο κριτήριο που χρησιμοποιείται για να επιλεχθούν οι θέσει εργασίας που θα χαθούν ε, είναι ε, εάν ο εργαζόμενος είναι εκείνος ο οποίος κερδίζει τα χρήματα για να συντηρήσει την οικογένειά του. Εκεί δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση φύλου. Επίσης, ο φορέας ο οποίος ασχολείται με την βία κατά των γυναικών δεν απασχολεί αρκετά άτομα. Δεν έχει αρκετό προσωπικό για να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Μάλιστα, σε ορισμένε περιπτώσεις, ε, αρχές, οι οργανισμοί οι οποίοι ε, ε, είχαν ως θέμα την προστασία των γυναικών καταργήθηκαν ή ενσωματώθηκαν και χάθηκαν μέσα σε μεγαλύτερους οργανισμούς και φορείς όσοι οργανισμοί και ιδρύματα έχουν ως στόχο την, τον αγώνα της επιβολής της ισότητος υπέρ των γυναικών θα πρέπει να ακούγονται, θα πρέπει να, έχουν, να είναι ισχυροί και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου κρίσεως. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν να επενδύσουμε σε αυτούς τους φορείς, σε αυτούς τους οργανισμούς και πρέπει να αναφερθούμε, να εστιάζουμε την προσοχή μας συνέχεια στην συμμετοχή των γυναικών σε οικονομικές δραστηριότητες. Παραδείγματο χάρη, να τις βοηθούμε, να τις υποστηρίζουμε και ενισχύουμε στην παροχή δανείων, στην, ε, σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης, στη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στις γυναίκες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση ε, διαφόρων, ε, ε, ας πούμε, εναλλακτικών μορφών ενέργειας για οικιακή χρήση, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να το εκμεταλλευτούν. Δεν ξέρω πότε είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Αλλά πιστεύω ότι και τον Απρίλιο θα μπορέσουμε στην επόμενη συζήτηση να ενσωματώσουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πλούμη, κυρία Κουρμάη. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα κι εγώ, κι εγώ να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που είπαν ότι χρειαζόμαστε θετική διάκριση υπέρ των γυναικών για να δούμε περισσότερες γυναίκες σε ισχυρές θέσεις, σε ηγετικές θέσεις. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια πρόταση να να κάνουμε μια έκθεση για την ισότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να μας υποστηρίξει. Στην προηγούμενη θητεία δεν μας υποστήριξε. Συνάντησα, ε, ε συμμετείχα στο hearing ε, που, που έγινε του κυρίου Βόζα Κότσιν και ευχαριστώ ιδιαίτερα τη γραμματεία που προετοίμασε αυτή την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό ο εισηγητής, ο κύριος Δρομέβα, που εργάστηκε από αυτού του θέματος πολύ καιρό, να εστιάσει πάνω στα βασικά θέματα και να επιφέρει μία ε, ισορροπία τις διάφορες ε, πτυχές της έκθεσης. Πρέπει επίσης ε, να αναφέρει ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετική προσέγγιση, διαφορετική ερμηνεία του τι σημαίνει κίνδυνος, ε, η αξιολόγηση του κινδύνου, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες είναι αυτές που λαμβάνουν αποφάσεις. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε περισσότερο την πλευρά των πολιτών μας. Εμείς οι γυναίκες συνήθως παίρνουμε μία απόφαση σύντομα, λέμε ένα, δύο, τρία και την παίρνουμε την απόφαση και συνήθως είναι και μακροχρόνια η προοπτική την οποία ε, αντιμετωπίζουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κατασκευαστικός ε, τομέας είναι αυτός ο οποίος εθίγει περισσότερο από την κρίση και περισσότεροι εργαζόμενοι ήταν άντρες σε αυτό το τομέα. Και οι πάρα πολλές τράπεζες χρεοκόπησαν, αλλά δύο-τρεις τράπεζες επιβίωσαν επιτυχώς και μάλιστα σε μία τράπεζα η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν γυναίκες και αυτή η τράπεζα επιβίωσε. Πρέπει λοιπόν ε, να κλείσουμε και το χάσμα που υπάρχει ε, στις αμοιβέ το 2007 γιορτάσουμε την 50η επέτειο της συνθήκης της Ρώμης, η οποία ήδη από τότε, μισό αιώνα πριν, είχε θεσμοθετήσει ίση αμοιβή για ίση εργασία. Σας θυμίζω λοιπόν ότι η έκθεση λέει ότι αν συνεχίζουν τα πράγματα ως έχουν θα χρειαστούμε 70 χρόνια για να κλείσει αυτό, αυτό το χάσμα, για να γεφυρώσουμε τη διαφορά των αμοιβών. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και ήδη ελέγχθη ότι το 2010 πρέπει να μια γυναίκα να εργαστεί 60 μέρες περισσότερο για να μπορέσει να πάρει την ίδια αμοιβή. Δεν είναι μόνο όμως ε, δύο μήνες, ό,τι περισσότερα παιδιά έχεις, ε, τόσο ε, περισσότερο διάκριση υφίστασε και τόσο πιο δύσκολα είναι να επιτύχεις την ισότητα. Μπορεί να χρειαστεί τρεις-τέσσερις μήνες παραπάνω να εργαστεί για η διαμοιβή. Λοιπόν, πολλά τέτοια θέματα υπάρχουν και ισχύουν και ας μην ξεχνάμε και τις στατιστικές του Eurostat για τη διάσταση του φιλού. Εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί πρέπει να επιβάλλουμε την ε, πολιτική μας βούληση. Πιστεύω ότι η Επιτροπή μας έχει αυτή τη βούληση και εγώ υποστηρίζω την έκθεση ολόψυχα και συγχαίρω τον εισηγητή. Ευχαριστούμε κυρία Γκουρνάη, κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, κάπως με εκπλήσει το πόσο αρνητικό είναι το, το κλίμα για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Πολύ φλού. Είναι τα πράγματα και επιπλέον ε, βλέπει, παραβλέπει άδειο το, το, το ποτήρι, μισοάδιο τέλος πάντων η συγκήτρια. Γιατί πάρα πολύ βασικοί οικονομολόγοι λένε ότι η συρρήγνωση του πιστοτικού τομέα είναι ε, μια καταστροφή που προκλήθηκε από άντρες, γιατί είναι τόσοι πολλοί άντρες που είχαν ταινίε σε αυτόν τον τομέα. Αλλά εγώ νομίζω ότι ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου κατηγορίε. Θα πρέπει να λέμε ότι το σύνολο, το σύνολο του κλάδου δεν θα έπρεπε να περιορίζει την πίστη, την δανειοδότηση. Αλλά γιατί τώρα να δαιμονοποιούμε τους άντρες. Σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι κάποια μέτρα υπέρ της ισότητας ματαιώθηκαν ή καθυστέρησαν. Εγώ στη χώρα μου δεν είδα τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Γιατί να λέμε τέτοια πράγματα. Είναι βάσιμα. Ας πούμε εκεί που λέει ότι υπάρχει πέρα μια μεταλλαγή και περιθωριοποίηση λόγω της οικονομικής κρίσης. Τι είναι, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά. Θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το κείμενο για να μην καταλήγουμε σε τέτοια γελιοποίηση. Με τέτοιες ε, και χαρακτηρισμού. Επίση, παραπονιόμαστε ότι έχει υπερβολικά πολλέ γυναίκε στον δημόσιο τομέα. Ναι, αλλά. Ξέρετε. Ε, Όλε αυτέ οι γυναίκε στο δημόσιο που τα περνάνε πολύ καλύτερα από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον στη χώρα μου. και πρόκειται να πληρώσουν την ύφη όσον αφορά τις περικοπές του γενικής πρόνοιας κλπ. Έχουν γίνει σε κάποιες χώρες και θα πρέπει να γίνουν τέτοιες περικοπές. Και λέγεται το κυρίω οι γυναίκε την πλώσουν τη νύφη, όμω εγώ επαναλαμβάνω ότι ούτε δυσμενή διάκριση υπάρχει στη χώρα μου στι γυναίκε στο δημόσιο ούτε μισθολογική διάκριση άλλου είδου ε, και όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασία. Οι άντρε υφίστανται δυσμενή διάκριση στην, στον τομέα τη παιδεία, γιατί εκεί έχει ιδιαίτερα πολλέ γυναίκε. Και εν υπάρχει μισθολογική ισότητα στον κλάδο αυτό. Να το δούμε πιο θετικά, να δούμε πιο πολλούς άντρες και σε θέσεις δασκάλων, καθηγητών. Να δούμε πώς θα έχουμε πιο πολλούς δικαστές άντρες. Γιατί είναι συντριπτική πλειοψηφία των ε, γυναικών που έχουν τις δικαστικές θέσεις ε, άλλωστε έχουν σπουδές πάρα από αυτές ε, νομικά, οπότε ε, είναι πιο καλά εξοπλισμένες σε αυτές τις ε, θέσεις του δημόσιου τομέα, κυρίως εκεί παρά όσον αφορά τον ανοίξουν ένα Άρα προσοχή, προσοχή για τέτοιου είδου κρίσεις. Τώρα, παρακάτω. Μετανάστες. στη χώρα μου, αυτοί οι μετανάστες ως εργαζόμενοι έχουν ε, την ίδια προσβασιμότητα στην υγεία, τα ίδια δικαιώματα. Γιατί λέμε τέτοια πράγματα εδώ, ότι υπάρχει περιθωριοποίηση των ε, μεταναστών, ναι, των λάθρων μεταναστών, όχι των νομίμων μεταναστών. Και άλλα, και άλλα μπορούσα να σας πω από το κείμενο. Άρα, Πού το πάω. Θα πρέπει να προσέξουμε τι λέμε. Ποιον, τι καταδικάζουμε. Μην γενικολογούμε. Επίσης έχουμε για την διάθεση παρελθόν 20 σε επιφυλάξεις ε, σε σχέση με τα 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πράσινες. Επίσης, υπάρχει μισθολογική ανισότητα. Παντού. μου για το περίφημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την ημέρα της γυναίκας και εκεί για αυτή τη χάρτα που λέω ότι πρόκειται να γίνει αυτή η προσπάθεια με ορίζοντα το 2014. Έχουμε και αυτή την οδηγία. Το 75, 35 χρόνια υπάρχει αυτή η οδηγία. Ποια αναρωτιέμαι. Με ποια μέτρα. Με ποια μέσα πολιτικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει ούτως ώστε να κάνει τη δουλειά της και να μπορέσει να εφαρμόσει ορθά αυτήν την οδηγία που είναι πάρα πολύ αξιόλογη μια που στην ε, χώρα μου ε, πάρα πολλές γυναίκες έχουν ωφεληθεί στο δημοσιο τομέα. Γιατί προσέφηκαν δυνάμει αυτής της ε, οδηγίε είχαν το θάρρος να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους και έχοντας στο χέρι αυτήν τόσο αξιόλογη οδηγία. Οπότε υπάρχει αυτό το μισθωτικό χάσμα, λένε σαφέ ότι αυτό αφορά κάποιους οικονομικούς κλάδου δραστηριότητα. Σε κάποιου οι γυναίκες κυριαρχούν, σε άλλους κλάδους το χάσμα αυτό είναι πολύ πιο μικρό από άλλους. Έχουμε τα συνδικάτα, τους κοινωνικούς εταίρους που προχωρούν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και ε, θα ξέρω ακριβώ τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το μέσο του 2014 για τη μείωση του χάσματο στη Γερμανία. Το ΑΕΠ λέει ότι αν γυρθεί αυτό το χάσμα θα έχουμε 30% αύξηση του ΑΕΠ. Μα ποιος κάθισε και το υπολόγισε αυτό. Δεν είναι αυτό μια υπερβολή. Μα αν ήταν έτσι τότε μαγικά θα εξαφανιζόντουσαν τα, τα πράγματα. Δεν θα είχαμε πρόβλημα ανάπτυξη στην οικονομία μας εάν ίσχυε κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είναι τα σενάρια τόσο εύκολα όσο αναφέρονται εδώ. Και εδώ είναι αναφορά σε αυτή την περίφημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, να λέμε πως την ανακοίνωση της Επιτροπής και να μην προβαίνουμε σε τέτοιου μεγαλόστομες διατυπώσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Λίλη. Να ρωτήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής αν θέλουν να λάβουν το λόγο. Ε, να δώσω λοιπόν το λόγο πάλι στον εισηγητή. Έγινε αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και με τις τροπολογίες θα μπορέσουμε να επιφέρουμε κάποιες διορθώσεις, κάποια πράγματα να διευκρινιστούν, κάποια στοιχεία τα οποία δεν τα έχει η αρχική εκδοχή του κειμένου. Για να δούμε τι δεν αναφέραμε ή τι δεν τονίσαμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία τα, το τόνισε η κυρία Μωρέν Σορτιέ αλλά και η κυρία Λούλινγκ. Αυτό που θα σας πω αφορά την βία κατά των γυναικών. Κάτι το οποίο έχει παροξενθεί. Είναι φαινόμενο που στατιστικά φαίνεται ότι παροξύνεται σε περίοδους κρίσης λόγω έλλειψης ασφάλειας, απώλεια ε, δουλειάς και μας οδηγεί μέσα σε κάποιες βίες εκδηλώσεις των οποίων θύματα κυρίως είναι οι γυναίκες. Πρόκειται επομένως για δυσάρεστη συνέπεια των άστοχων πολιτικών που ακολουθήσαμε. Να μην υπόψη τι γίνεται στις περιπτώσεις που η γυναίκα είναι ο μόνος που εργάζεται. Ποιες είναι οι συνέπειες του όταν μια τέτοια γυναίκα χάσει τη δουλειά της. Από αυτά που άκουσα, πάντως, στέκομαι στα εξή. Πρώτον, συμφωνώ και είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται να δώσει το καλό παράδειγμα το δημόσιο, κυρία Μωρέν Σορτιέ. Είναι πολύ σημαντικό. Και όταν κάτι ζητούμε από τον ιδιωτικό τομέα, τότε το ίδιο πράγμα θα πρέπει πρώτος να το κάνει δημόσιος τομέας. Ούτε να ξεχνούμε ότι και ο προϋπολογισμός και η απασχόληση στο δημόσιο και η φορολογική πολιτική, όλα αυτά επιδέχονται διόρθωση από πλευράς των φύλων. Και επομένως μέσω αυτών των πολιτικών Μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις αδικίες, τις ανισότητες που υπάρχουν στην κοινωνία και δεν γίνονται αλλιώ. Λέμε τώρα, το πώς θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε κάποια μέτρα. Πώς θα διευκολύνουμε την ένταξη των γυναικών σε κάποιες υπεύθυνε θέσεις, σε θέσεις λήψης αποφάσεων, κάτι το οποίο ανέκαθεν πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε τέτοια μέτρα όχι σαν μοναδικά μέτρα, αλλά σαν τμήμα του προστασίου μέσω του οποίου θα προχωρήσουμε σε κάποιες πολιτικές. Τώρα για τη συνεννόηση, συμφιλίωση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν έχουμε τροπολογίε, θα πρέπει να γίνουν. Στο, στο αντίστοιχο σημείο του και δεν μιλώ για συνεννόηση, συμφιλίωση ε, σε επίπεδο επαγγελματικό ή οικογενειακό. Μιλώ για το τι γίνεται σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο ανάπτυξης προσωπικότητας. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από τις οικογενειακές ευθύνες που τυχόν έχει κανείς. Τελευταία μου σκέψη, με αφορμή τα όσα μας είπε η κυρία Λούλινγκ. εγώ δεν έβγαλα τίποτα από το κεφάλι μου. Όλα αυτά έχουν ως πηγή το δημόσιο. Είναι κρατικές πληροφορίες. Αλλά θα πω όλοι μπορούν να τα γνωρίζουν. είναι στοιχεία που τα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, α πούμε στη, διάταξη 20, σε σχέση με την οικολογική πολιτική, όπως είπε η κυρία Λούλινγκ. Μπορεί κανεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, αλλά τα στοιχεία αυτά είναι, είναι δεδομένα. Αφού λέμε για τέτοιες πηγές πληροφοριών, πώς αμφισβητούνται. και εκεί που αναφερόμαστε και είπε και η κυρία Λούλιν για την υποχρέωση της γυναίκας να διεκδικεί τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 δεν είναι η Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στις άλλες χώρες. Θα πρέπει όλα αυτά να τα βλέπουμε στο πανενωσιακό πλαίσιο. Φυσικά και κάποιες χώρες είναι παράδειγμα προς ε, μίμηση. Αλλά να μην ξεχνούμε την Ευρώπη των 27, όπου σε κάποιες χώρες είναι διαφορετικά τα πράγματα, οπότε και επιβάλλεται να γίνουν κάποιες πολιτικές, να ληφθούν κάποια μέτρα που δεν χρειάζονται αλλού. Έτσι, επομένως, θα πρέπει να αντικρίζουμε την ενωσιακή πραγματικότητα. Πάντως, απλώς εδώ λέμε για κάποια ε, αφετηρία που αποτελεί αυτό το κείμενο. Θα μελετηθούν οι τροπολογίες με καλή θέληση, με προσοχή και το θέμα δεν είναι τι θεωρείται αξιόπιστο, τι πιστεύει κανείς, αλλά το τι μπορεί να είναι χρήσιμο. Πρόεδρος. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τους συναδέλφους για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. 23 Μαρτίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε 3-4 Μαΐου και στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ όλους και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε για το επόμενο θέμα 7. είναι η των αποτελεσμάτων του χάρτη πορείας 2006-2010 για την ισότητα και συστάσεις για το μέλλον. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον για αυτό το θέμα. Και η συγγήτρια είναι η κυρία Φιγκουερέδο από την ΚΟΕ και στην συνεδρίαση του Οκτωβρίου είπαμε ότι είναι σημαντικό να συμμετάσχουμε σε αυτό το θέμα με μία έκθεση και το ανασέσαμε στην κυρία Φιγκουερέδο. Αυτό το που νομίζω πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ζητήσουμε από την εισηγήτρια να μας ενημερώσει και μετά θα διεξαγάγουμε τη συζήτηση και θα συζητήσουμε την... θα εξετάσουμε την έκθεση, το σχέδιο έκθεση. Δίνω στην εισηγήτρια το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή, όπως ε, αναφέρατε στόχο έχει να παρουσιάσει ένα σύνολο προτάσεων τις οποίες θα μπορούσε να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την εκπόνηση της νέας στρατηγικής για την ισότητα. Όλα αυτά κατόπιν της σχετικής συζήτησης που είχαμε εδώ. Όμως στο μεσοδιάστημα είχαμε και άλλες διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με την Επίτροπο Ρέντινγκ και μας δόθηκε η πληροφορία ότι προτίθεται να μας ακούσει για να λάβει πράγματι υπόψη τις θέσεις των μελών αυτής της Επιτροπής και για να υποβληθεί τελικά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο της φετινής χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο χρόνο από ό,τι αρχικά προβλέπαμε. Νομίζαμε ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο και μας πίεζε κάπως ε, το χρονικό περιθώριο για να συνεισφέρουμε στη νέα στρατηγική. Όμως μετά τις συνομιλίες μας με την κυρία Ρέντινγκ και Πρόεδρε, και εσεί γνωρίζετε την πληροφορία αυτή από το πρωινό τη περασμένης εβδομάδας. Υπάρχει δέσμευση για διάλογο μαζί μας για το θέμα αυτό και ε, η εργασία αυτή θα γίνει από κοινού ώστε να σχεδιάσουμε κάποια σημαντικά βήματα και να μην παραμένουμε σε μια απλή δήλωση προθέσεων όπως και έγινε με τη χάρτα. Τώρα θέλουμε να περάσουμε στην πράξη, να κάνουμε πραγματικότητα, να υλοποιήσουμε όσα προβλέπει η στρατηγική για την ισότητα. Άρα, και εφόσον το κείμενο αυτό το έχουμε ετοιμάσει ήδη πριν από τις τελευταίες εξελίξεις, σε κάθε περίπτωση Όταν είδαμε το χάρτη πορείας ε, για την ισότητα 2006-2010 και τον εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ότι κάποια δεδομένα ξεχωρίζουν και είναι κάποιες σημαντικές πτυχές ε, της ισότητας μεταξύ, ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που θα πρέπει να τονίσουμε. Όμως δεν είναι ανάγκη να τα επαναλάβουμε, τα έχουμε ξανασυζητήσει, έχουμε επισημάνει τις ελλείψεις, λίγη πρόοδος επιτελέστηκε, υπήρξαν και κάποιες το στοχωρήσει. Νομίζω τώρα το σημαντικότερο είναι να σκεφτούμε τι οφείλουμε να κάνουμε για να υπάρξει ένα πραγματικό άλμα σε αυτή την διαδικασία. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι ένα μεγάλο βήμα θα πρέπει να γίνει και στο πολιτικό πεδίο. Δηλαδή, δεν έχουμε πλέον ένα απλό χάρτη πορείας ούτε μια απλή πρόθεση δηλώση, δήλωση προθέσεων. Έχουμε κάτι πιο δεσμευτικό, πιο ισχυρό. Γι' αυτό η έκθεση που έχω υποβάλει χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα στο θεσμικό κεφάλαιο με μια σειρά από προτάσεις και το άλλο στους στόχους, κεφάλαιο που καλύπτει τους στόχους. Όπως τα γνωρίζετε έχουμε κάποια όρια στο πόσους χαρακτήρες μπορεί να περιλαμβάνει η έκθεση σε αυτή την προκατακτική φάση και ευχαριστώ εδώ και την γραμματεία της Επιτροπής για τη στήριξη που μας έδωσε. Ίσως η έκθεση ξεπερνάει κάπως ήδη τα περιθώρια, όμως ε, είμαστε ακόμα στην προκαταρκτική φάση, μετά θα περάσουμε στις τροπολογίες και τις αλλαγές είτε από μένα την ίδια είτε από τους συναδέλφους, οπότε θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Πάντως, στο θεσμικό επίπεδο, ποιε είναι οι βασικές προτάσεις που περιλαμβάνονται εδώ. Από τη μια, να έχουμε μια ημερήσια διάταξη για δράση και πολιτικούς συμβιβασμούς βάσει της πλατφόρμας του Πεκίνου, και τονίζοντας πάντοτε τη σημασία της συμβολής του Συμβουλίου που θα πρέπει να εγκρίνει τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να μην είναι αυτή μια πρόταση απλώς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γιατί, διότι έχουμε τη στρατηγική 2020 πρόταση της Επιτροπής που όμως θα κυρωθεί και από το Συμβούλιο. Και για τις γυναίκες αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ. Άρα θα πρέπει να γίνει ένα πολιτικό άλμα εδώ στην όλη διαδικασία. Να υπάρξει μια δέσμευση, ανάληψη ευθυνών και από τους κυβερνήσεις, από τα κράτη-μέλη. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν ένα βήμα σημαντικότατο. Προφανώς μετά θα έχουμε και την ε, τοποθέτηση του Ευρωκοινοβουλίου για να διασφαλίσουμε αυτή τη νέα όθηση στην πολιτική της ισότητας. Έπειτα θα πρέπει συστηματικά να παρακολουθούμε την, ε, πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες. Όχι μόνο μια φορά την πενταετία, αλλά κάθε χρόνο κάποιες δράσεις να υλοποιούνται, ώστε να υπάρχει πραγματική παρακολούθηση ε, στην πράξη και πολιτική της όλης διαδικασίας. Δηλαδή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να δημιουργήσουν κάποιου είδους τριμερούς τακτικής συνάντησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για να παρακολουθούμε την πρόοδο της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κάθε χρόνο θα πρέπει να οργανώνεται αυτό, είτε τον Οκτώβριο, είτε στο τέλος του χρόνου, είτε στην αρχή της χρονιάς, όμως κάθε χρόνο θα πρέπει να υπάρχει αυτή η χρονική, αυτό το ραντεβού, αυτή η συνάντηση. Και θα πρέπει όλοι να αναλάβουν την ευθύνη για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Από την άλλη, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να προβάλλουμε περισσότερο όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν και τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες, τις γυναίκες, οι οποίες θα πρέπει να συμμετέχουν μέσω των ενώσεων, των ε, οργανώσεών τους, μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεων των κρατών μελών, αλλά και τα μέλη των διαφόρων εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών. Βεβαίω, πέραν των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πιστεύω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη προβολή, να ε, δοθεί έμφαση σε όλο αυτό το έργο. Να θυμίσω εδώ ότι στο Ευρωκοινοβούλιο στα πλαίσια της θετικής της Λισαβόνας υπήρχε κάθε χρόνο κάτι για την ισότητα των φύλων. Όμως το θέματα των γυναικών ουδέποτε έλαβαν την προσοχή που τους άξιζε ή τόσο πολύ προσοχή. Πιστεύω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα ενώπιον των δυσκολιών που έχουμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε την απαραίτητη όθηση, να κάνουμε τα θετικά βήματα που απαιτούνται Πρέπει να αξιοποιήσουμε τέτοιους μηχανισμούς που προϋπάρχουν από άλλους τομείς, να τους χρησιμοποιήσουμε και για την πολιτική της ισότητας των δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προφανώς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα εννοείται εφόσον θα αρχίσει πλήρως να λειτουργεί από τον Ιούνιο, θα δώσει κάποια αποτελέσματα. Πιστεύω όμως ότι εντωμεταξύ πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση να είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά πράγματι λειτουργούν, ότι υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα, γιατί μετατίθεται ένα άλλο πρόβλημα. Η πολιτική ισότητα απαιτεί και χρήμα, κονδύλια. Δεν μπορεί να είμαστε πάντα φτωχοί συγγενεί του προαπολογισμού και εδώ δεν μιλώ μόνο για το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και για το ευρωπαϊκό μαζί με το εθνικό. Είμαστε πάντοτε ο φτωχό ο συγγενή. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε Επίσης, σήμερα ασκείται σοβαρή πίεση και καλώς ώστε οι πολιτικές αυτές που, για τις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο να αναλύονται, από, να, να είναι αντικείμενο μελέτης αντικτύπου από κοινωνικής άποψης. Συμφωνώ, πρέπει να υπάρχει όμως ανάλυση και του αντικτύπου στην πολιτική της ισότητας ποιε είναι οι συνέπειε για τι γυναίκε από τι διάφορε πολιτικέ αποφάσει. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα έχουμε μία διαρκή πίεση ώστε επιτέλους το θέμα αυτό να αποτελέσει ζήτημα των καθημερινών συζητήσεων των πολιτικών ευθυνόντων, των αρμοδίων, των όσων λαμβάνουν αποφάσεις στο ευρωπαϊκό, περιφερειακό, τοπικό, εθνικό επίπεδο, σε όλα τα κλιμάκια. Γι' αυτό πιστεύω ότι στην πράξη η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις γενικές της κατευθυντήριες γραμμές, προτάσεις που ούτως ή αναφέρονται στην γνωμοδότηση, πρέπει να δημιουργήσει μηχανισμούς διαρκούς παρακολούθησης και υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα και την ισότητα των δικαιωμάτων. Ίσως να μας πούνε ότι κάποια στοιχεία προϋπάρχουν. Εγώ νομίζω όμως ότι ο πραγματικός συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών συνιστοσών και των υπηρεσιών δεν λειτουργεί προφανώ αρκετά αποτελεσματικά. Υπάρχουν αντιπαραθέσει και αντιφάσει συνεχώ στην πράξη και το διαπιστώνουμε καθημερινά. Επίση, είναι σημαντική είναι σημαντικό η πολιτική αυτή να καλύπτει διαφορετικούς τομείς. Τον οικονομικό. Μόλις τώρα ακούσαμε τον συναδελφό μας να μας αναπτύσσει τα σχετικά επιχειρήματα. Τον κύριο Ρωμέβα με την εκθεσή του. Στον οικονομικό τομέα, τον χρηματοπιστωτικό, τον κοινωνικό, του προπολογισμού. Θα πρέπει να αναζητήσουμε μια προσέγγιση που όμως να γίνει πραγματικότητα. Όλοι συμφωνούν ότι η πολιτική ισότητα πρέπει να υλοποιηθεί, αλλά πολλές φορές αυτά παραμένουν μόνο λόγια στο χαρτί. Και όταν έρχεται η ώρα να υλοποιηθούν, κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Ήρθε λοιπόν η ώρα να γίνουν όλα αυτά πράξη. Επίσης, η διάδοση των παραδειγμάτων καλών πρακτικών, η πραγματική παρακολούθηση των όσων συμβαίνουν και η διάδοση των καλών παραδειγμάτων, εδώ μπορεί να διδραματίσει ρόλο η Επιτροπή μας, εμείς οι ίδιοι που γνωρίζουμε τα καλά παραδείγματα να τα διαδώσουμε, αλλά και η Εκτελεστική Επιτροπή να φροντίσει για τη διάδοση των πρακτικών των κρατών μελών διότι αυτό θα έχει νόημα και για τους υπόλοιπους. Επίσης, πρέπει να επιμείνουμε στην διτή προσέγγιση. Μια στρατηγική που να επιτρέπει από τη μια την ενιαία προσέγγιση του θέματος της ισότητας των φύλων, αλλά ταυτόχρονα να μην παραμελούμε τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται. Να συμπεριλαμβάνονται νομοθετικά μέτρα, μέτρα στον προϋπολογισμό, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πολιτικής της ισότητας είναι η έλλειψη ακριβώς παρακολούθησης, ελέγχου της υλοποίησης. Εδώ χρειάζεται να συζητήσουμε ξανά και ξανά και με τα κράτη-μέλη μαζί διότι αυτό δεν το λέω γιατί θέλω να επιβληθούν κυρώσει στα κράτη-μέλη. Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κάποιο κράτο μέλο. Αλλά υπερασπίζουμε εδώ την περισσότερη ανάληψη ευθυνών από όλε τι πλευρέ. Υπάρχουν διαφορετικέ προτάσει και μέτρα που μπορούν να αναλυθούν στο θεσμικό επίπεδο, ώστε οι πρακτικέ ετησίω να ελέγχονται, να ενημερώνονται, να διαδίδονται για το τι γίνεται. Και να υπάρχουν έπειτα και μέτρα κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση μέσω τη διάδοση των καλών πρακτικών να δοθούν ενδεχομένως βραβεία για διάφορα θέματα, σε διάφορους τομείς, για όσους διακριθούν σε κάτι, για όσους καταφέρουν να επιτύχουν περισσότερους στόχους, περισσότερα αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνουν όλα αυτά χωρίς να αναλάβουμε μέτρα τιμωρητικά. Δεν υπερασπίζομαι κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι εδώ ακριβώς, το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις διάφορες αντιπροσωπίες εδώ οι ίδιες εμείς στην Επιτροπή μας, ως μέλη αυτής της Επιτροπής, <clears throat> πρέπει να συζητούμε πώς στις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου και στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα της ισότητας, να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου μέσω όμως της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους συναδέλφους μας, τις συναδέλφους μας, όλους όσους συμμετέχουν σε αποστολές και αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου. Αυτό στο πολιτικό επίπεδο από θεσμικής άποψης και πολιτικής άποψης είναι απαραίτητο να γίνει. Έπειτα προφανώς υπάρχουν και οι στόχοι. Στους στόχους προφανώς είναι σοβαρό το έργο που ήδη γίνεται. Νομίζω ότι η Σουηδική Προεδρία έκανε πολλά ενδιαφέροντα, μεταξύ των οποίων το βιβλίο που δημοσίευσε για την ανάλυση της πλατφόρμας του Πεκίνου ΣΥΝ 15. Αυτή ήταν μια αξιόλογη συμβολή, όμως θα πρέπει το έργο αυτό να συνεχιστεί να αναπτύξουμε τους κατάλληλους δείκτες, να έχουμε στόχους, να υιοθετήσουμε τις απαραίτητες πολιτικές στους 12 τομείς που προβλέπονται. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη σε αυτή τη φάση έχει μια πολύ καλή βάση εργασίας, ώστε να συνεχίσει, να εξακολουθήσει και να δώσει κίνητρα ώστε να βελτιωθεί αυτή η βάση εργασίας εξ αφορμής των όσων ήδη έχουν γίνει. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει χειραφέτηση των γυναικών εάν δεν ανεξαρτοποιηθούν οικονομικά. Η καταπολέμηση της φτώχειας έχει πολλές φορές γυναικείο πρόσωπο. Ιδού γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε την κακοπληρωμένη εργασία, την προσωρινή εργασία, την ανεργία. Είναι σημαντικό να δώσουμε, να κινητοποιήσουμε και τις υπόλοιπες πολιτικές ε, στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Ιδίω σε μια φάση όπως η τωρινή, όπου σχεδιάζονται και λαμβάνονται αποφάσεις που επιβαρύνουν τη θέση των γυναικών. Επιβαρύνουν κάποιες φορές τις δυσκολίες τους, δυσχεραίνουν ε, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες τις οποίες ζουν και επιτείνουν τη φτώχεια τους. Εδώ λοιπόν χρειάζονται ισχυροί, σοβαροί στόχοι. Και στην πράξη θα πρέπει να έχουμε πολιτικές που να δίνουν κίνητρα για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες, βασικά για τις γυναίκες, όπως τον κοινωνικό τομέα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε το θέμα της παραγωγής, τη διάσταση των ε, κρατικών δημοσίων υπηρεσιών ποιότητα. Διότι ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε προβλήματα των πληθυσμών, αλλά ειδικώ των γυναικών σε διάφορα επίπεδα. Δίνοντα δουλειά, θα του τους βοηθήσουμε να καταπολεμήσουν την φτώχεια. Σε ό,τι αφορά την διακριτική μεταχείριση και τι διακρίσει, ήδη κάποιε προτάσει πρέπει να ληφθούν υπόψη, διότι γνωρίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις γίνονται ενδιαφέρουσες προσπάθειες, αλλά κάποιες φορές γίνονται και αντιφατικές κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη. Ε, πρέπει οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται για την ισότητα των φύλων, για την ισότητα μεταχείριση της επιχειρήσης, να συνδυαστούν με άλλες πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα Equal δεν αρκεί η συνέχεια του προγράμματος δεν έδωσαν τα αποτελέσματα τα αναμενόμενα. Τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες που εγώ γνωρίζω καλά. Υπήρξαν λοιπόν αντιφατικότατες πολιτικές και αυτό πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Τι θετικό έχει γίνει και πιθανώς να ξαναδούμε και να διορθώσουμε αυτά που δεν ήταν τόσο θετικά. Προφανώς οι πολιτικές ευαισθητοποίησης, η φορολόγηση ε, της εργασίας είναι καθοριστική σημασίας. Στην χώρα μου, όταν μιλώ με γυναίκες, ακούω συνήθως τις ίδιες κριτικές ε, για τις επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση που πάλι προέβλεψε ένα βραβείο και δεν το έδωσε σε αυτόν που μπορεί να το άξιζε γιατί μπορεί να απουσίαζε για να πάει το παιδί του στο γιατρό, γιατί είχε κάποιο ιατρικό ραντεβού και πολλές φορές οι γυναίκες που αξίζαν τα βραβεία αυτά, τα, την επιβράβευση αυτή για την εργασία τους τελικά δεν την έλαβαν ποτέ και αυτά τα 50-100 ευρώ τα χρειάζονται πραγματικά για την καθημερινή του ζωή. Άρα η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται, οι προμοδοτήσεις δεν δίνονται πάντοτε. Εδώ πρέπει να απαιτήσουμε σε επίπεδο 100 μελών να ληφθούν μέτρα, να εμποδίζουν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες αδικίες αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και διαρκές, διαρκείς μορφές ε, παρέμβασης στην πράξη. Εδώ θα συμφωνήσω με κάποιους συναδέλφους που λένε ενίοτε ότι είναι σημαντικό να δίνουμε προσοχή στην υλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσία. Δεν θέλω βεβαίως με αυτό να πω ότι δεν χρειάζεται να πάμε και παραπέρα, εφόσον είναι δυνατό. Όμως πρέπει να επιμείνουμε στην υλοποίηση των υπαρχόντων νομοθετημάτων. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες πτυχές που έχουμε κατά καιρό συζητήσει εδώ, όπως κάποια από τα τελευταία ζητήματα που μας απασχολήσαν με εκθέσεις, τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, όπως εκείνες που φέτος ήδη έχουμε συζητήσει, για την ε, καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων, για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τελευταία έκθεση του κ. Ταραμπέλα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που μαζί με το ψήφισμα που κάναμε για τη διάσκεψη του ΟΗΕ είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά να τα δώσουμε στην Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος της συνεισφοράς μας για τη νέα στρατηγική της ισότητας και στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησής μας. Συνάδελφοι, αυτά είχα να σας πω προς στιγμή για το θέμα αυτό. Είμαι ανοιχτή βεβαίως σε όλες τις προτάσεις, συμβολές που μπορεί να υποβάλλετε, τις ιδέες που μπορεί να έχετε. και είμαι έτοιμη να τα συζητήσω με όλους τους συναδέλφους όλων των πολιτικών παρατάξεων. Ευχαριστώ κυρία Φιγουρέιντο για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση αυτής της σημαντικής έκθεσης και τώρα θα, δώσω, θα, κάνουμε, θα κάνουμε τη συζήτησή μας η κυρία Γκομάη καταρχάς. Ευχαριστώ αγαπητή πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, λίγη επαγγελματική εργασία και την ε, δέσμευση προς αυτό το θέμα της εισηγήτριας. Πριν από λίγο καιρό είχαμε συμμετάσχει σε στην σχετική ακρόαση και είχαμε ακούσει όλες αυτές τις ε, απόψεις και πιστεύω ότι μετά από την ακρόαση αυτή και από πλευρά τη κοινωνία των πολιτών ε, μπορούμε να ε, προβάλλουμε μια ισχυρή έκθεση. Θα ήθελα να προτείνω δύο ε, θέματα. Καταρχάς, στο σημείο 6 μιλάμε για την αξιολόγηση κοινωνικών θεμάτων. Εδώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τη διάσταση του φύλου γιατί εννοείται. Δεύτερον, πρέπει να τονίσουμε την τρέχουσα έλλειψη στατιστικών δικτών. Είναι απαραίτητο για να επιβάλλουμε ε, αποτελεσματικά την πολιτική της ισότητας πρέπει να έχουμε στατιστικά στοιχεία. Και ε, τρίτον ε, πρέπει να αναφερθεί όλος ο κύκλος της λήψης των αποφάσεων, δηλαδή υποβολή ενός προγράμματος, αξιολόγηση, απόφαση, εφαρμογή, υλοποίηση. Και αυτός είναι ο κλασικός κύκλος ε, ε, υλοποίησης ενός προγράμματος, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει χωρίς την απαραίτητη υποδομή. Το σχέδιο έκθεση. πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσει περισσότερο την ε, δεσμευτική νομοθεσία, ένα δεσμευτικό νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει να είναι δεσμευτικό και να διαθέσουμε τους απαραίτητους πόρους για να το καταστήσουμε δεσμευτικό. Και επίσης, όπως στο θέμα της βίας κατά των γυναικών, θα πρέπει να υπάρχει μία οδηγία ώστε η βάση όλης της τεκμηρίωσης να είναι νομικά δεσμευτική. Θα ήθελα να αναφέρω και ορισμένα άλλα, ορισμένες άλλες λεπτομέρειες που κρύβονται μέσα στο κείμενο, αλλά πρέπει να τονιστούν η διάσταση του προβλήματος πρέπει να τονιστεί. Είναι σημαντικό. Πρέπει να εξετάσουμε τα στοιχεία της απασχόλησης των γυναικών και των δεσμεύσεων του προϋπολογισμού ως προς τις γυναίκες. Και πρέπει επίσης να προβλέψουμε την στρατηγική εξόδου, ε, εξόδου από την αγορά εργασίας δηλαδή, που θα καλύπτει τις γυναίκες. Επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για την Ατζέντα 2020-2020. Η διάσταση ε, του φύλου στην Ατζέντα 2020 είναι εξαιρετικά σημαντική. Όπως είπε και η Κομισιόν, χρειαζόμαστε μια στρατηγική ε, ε, διάσταση των, φίλων φύλων στην Ευρώπη του 2020. Καλή είναι η ατζέντα της, Λισαβόνας, δεν πειράζει αν περιοριστούν ε, ορισμένοι στόχοι μας, αλλά ας επιβληθεί η διάσταση του φύλου στην Ατζέντα 2020. Στο νέο, στη νέα πορεία αυτή, στο νέο χάρτη πορείας ε, πρέπει να καλυφθούν όλοι οι αρμόδιοι οργανισμοί και φορείς και στην στρατηγική αυτή μεταξύ 2006-2010 είχαμε έξι σημεία τα οποία είχαμε αναφέρει γιατί προσθέσαμε και τις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση στις δικές μας απόψεις, διότι εμείς είμαστε το εκλεγμένο σώμα, εκλεγμένοι εκπρόσωποι και εμείς έχουμε επίσης τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με όλες τις μεγάλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με φορείς, ε, ε, γυναικείες οργανώσεις κλπ. Και γι' αυτό η στρατηγική μας ε, πρέπει να είναι στέρεη και δυνατή. Συμφωνώ επίσης και με την κυρία Λούλινγκ ότι αυτό το κείμενο το οποίο προετοιμάστηκε στη Νέα Υόρκη δεν είχαμε ακόμα τη δυνατότητα να το μελετήσουμε σε βάθος. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από όλες τις συναδέλφους μου και τους συναδέλφους μου η, κυρία Ρέντινγκ να, να έρθει να συζητήσουμε ε, διότι ξέρουμε ότι η Επίτροπος ε, είναι πρόθυμη να συνεργάζεται μαζί μας και να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φιγκερέρο ε, για την έκθεσή της. Είναι πολύ σημαντικό να συντάξουμε ένα, μια, έναν κατάλογο ενεργειών που πρέπει να κάνουμε. Το, λίγο το, το, φτιάξαμε αυτό με την έκθεση Ταραμπέλα που πέρασε από την Ολεομέλεια τον Ιανουάριο και πιστεύω ότι εδώ μια, υπάρχει μια προοδευτική πλειοψηφία με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και πιστεύω ότι αυτός ο χάρτης ε, πορείας θα δώσει την ευκαιρία να συνεργαστούμε ακόμα στενότερα. Όπως είπε, ε, η κυρία Ρέντινγκ δεν θα τροποποιήσει, δεν θα αλλάξει τη στρατηγική της, έχει παρουσιάσει τις ε, δεσμεύσεις της. Όπως είπαμε, αυτή, αυτός είναι ο χάρτης πορείας, τον οποίο πιστεύουμε ότι, τον οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε και να ενισχύσουμε. Ε, η κυρία Φιγκουερέιδο είπε ότι ήταν περιορισμένη όσον αφορά την, ε, τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της. Τώρα όμως μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε ώστε να ενισχύσουμε αυτή την αξιολόγηση. Υπάρχει βεβαίως καλά τεκμηρωμένα στοιχεία για την ε, ανισότητα στις αμοιβέ αλλά αυτό που δεν έχει καταγραφεί αποτελεσματικά είναι η φροντίδα και η περίθαλψη η οποία προσφέρεται από τις γυναίκες. Η συντριπτική πλειοψηφία των ε, ωφελούμενων από την περίθαλψη αυτή είναι άνδρες, αλλά και την, ε, τη φροντίδα αυτή την παρέχουν γυναίκες κατά, κατά πλειοψηφία. Αυτό δεν έχει καταγραφεί ακριβώς, αυτά τα ποσοστά. Επίσης ε, θέλουμε να συζητηθεί το θέμα της ε, δυνατότητας και της ε, της συμφιλίωσης της εργασίας με, τις, με τα εικονιακά καθήκοντα, με την εικονιακή ζωή και το θέμα των μειονοτήτων ε, που πολλές φορές αναγκάζονται να υφίστανται πολλαπλές ε, διακρίσεις ε, γυναίκες διαφορετικών εθνοτήτων που υποφέρουν από πολλές διακρίσεις. Επίσης το θέμα των λεσβίων γυναικών ή Um, των transsexuals που και αυτές οι ομάδες πληθυσμού υφίστανται διακρίσεις και πρέπει να καλυφθούν οι, οι ανάγκες αυτές νομικά ε, και να εμπίπτουν στο θέμα της διάκρισης ε, της διάστασης του φύλου και όχι του σεξουαλικού προσανατολισμού διότι οι διακρίσεις που υφίστανται αυτές οι ομάδες εμπίπτουν στη διάσταση του φύλου. Συμφωνώ γενικά με τις ε, ε, τον προσανατολισμό της κυρίας Φιγκουαρέιδο και πιστεύω ότι μπορούμε να τονίσουμε ακόμα ορισμένες πτυχές όπως αυτές τις οποίες ανέφερα για να ενισχύσουμε περισσότερο την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Λούλη. Euh, Θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε τι είδου ε, εκθέσει είναι αυτέ οι οποίε ε, κάνουμε εδώ. Γιατί εδώ πέρα διαπιστώνω ότι έχουμε την έκθεση. Ταραμπέλα, αυτό το σχέδιο τη έκθεση όσον αφορά την οικονομική κρίση και από την άλλη μεριά έχουμε και αυτό το σχέδιο της έκθεσης της κυρίας ε, Φιγερέντο που αφορά αυτό το χάρτη πορείας. Στις εκθέσεις αυτές επαναλαμβάνουμε αένα το ίδιο. Να μην γελιοποιηθούμε με αυτά τα πράγματα. Εγώ διαπιστώνω ότι εδώ υπάρχει ένα εδάφιο, μια παραγραφούλα που είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό το οποίο περιέχεται στην έκθεση Ταραβελά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα και στην έκθεση του κ. Ρουέδα, ε, όπως εδώ επομένως θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να γίνει, τι θέλουμε να υπάρχει το οποίο να μην είναι απαράδεκτο μια αποτελεί μια ακριβή επανάληψη, αντιγραφή. Ε, τα τελευταία 20 χρόνια ε, εγώ βλέπω τα ίδια να λέμε συνεχώς. Ε, μα είναι δυνατόν να δούμε πώς θα πούμε κάτι καινούργιο Όχι τα, τα ίδια, τις ίδιες γκρίνια, τις ίδιες γενικές διαπιστώσεις. Νομίζω ότι αυτό δεν αποτελεί αξιόλογο έργο ε, καμάρι της Επιτροπής μας. Είναι η τρίτη κατά σειρά έκθεση που τώρα λέμε ακριβώς τα ίδια. Και με καμαρών μου ότι κάναμε δήθεν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι έτσι δεν ε, μπορούμε να θεωρούμε ότι επιτελούμε νόμο παρασκευαστικό έργο σοβαρό. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κυρία Λούλιν για τις απόψεις σας. Τώρα ίσως το μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στην κυρίως συζήτηση. Ναι, κάποια πράγματα πρέπει να επαναλαμβάνονται, γι' αυτό επαναλαμβάνονται. Μέχρι ότου πετύχει κανείς το ότι επιδιώκει. Νομίζω ότι έχουμε εδώ πέρα κάποιε πάρα πολύ συγκεκριμένε προτάσει σχετικά με το πώ μπορεί να επιτευχθεί κάποια πρόοδο. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για να δούμε όμω τι άλλο θα μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν έχουμε εδώ πέρα βέβαια κάποιον την Επιτροπή που θέλει να λάβει το λόγο. Η θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Φιγκορέντο για να μας συνοψίσει και ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση απλώς θα σχολιάσω δύο από τις, παρεμβολ... από τις παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα για τις διάφορες προτάσεις και την ιεράρχησή τους. Προφανώς η Επιτροπή αυτή παίρνει πολύ σοβαρά το έργο της και γι' αυτό επαναλαμβάνουμε διαρκώς τις ίδιες προτάσεις για προβλήματα όμως που εμένουν εδώ και 20-30 χρόνια για τα οποία πρέπει να τα επιλύσουμε. Δεν έχουν βρεθεί λύσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή γίνονται προτάσεις ότι λύνονται και τα προβλήματα. Εάν τα προβλήματα εμένουν, πρέπει προτάσεις να ξαναγίνονται. Τι να κάνουμε, πρέπει η καταγγελία να παραμείνει. Δεν μπορεί να εξαλειφθεί, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε επειδή κουραστήκαμε λόγω κόπωσης. Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε τα είτε διότι όπως έχουμε πει τόσες φορές, κάποιες φορές ε, καλύτερο είναι να τηρούμε σιγή, Όμω όχι. Έτσι, όταν τα προβλήματα εμένουν, εγώ θα συνεχίσω λοιπόν. Και φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία των μέλων εδώ της Επιτροπής αυτήν την θέση θα προκρίνουν, θα προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών, τη ισότητα των φίλων, μέχρι να υλοποιηθούν τα ίσα δικαιώματα στην πράξη. Εδώ και 30-40 χρόνια μπορεί να χρειαστούν και 50 ή παραπάνω, αλλά θα συνεχίσουμε